Ας ξεκινήσουμε λοιπόν γιατί σήμερα έχουμε μια μεγάλη, ένα μεγάλο πρωινό με ψηφοφορίες. Και έτσι καλημέρα σε όλες και όλους πρώτα. Ξεκινάμε λοιπόν με το σημείο 14. Εκλογή του δεύτερου αντιπροέδρου λοιπόν. Έχουμε Έχουμε πρόταση της Γκουα. Η κυρία Μπιόρκ ζήτησε τον λόγο. Παρακαλώ, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Χαιρόμαστε που μπορούμε να παρουσιάσουμε την διάδοχο της Ίνες Ζουπέρ, ο Ζωάου Πουκμέντα Λόπες και θα θέλαμε να αναλάβει όλες τις αρμοδιότητες ε, της Ίνες ε, δέχτηκε. Θα ήθελα λοιπόν ε, να τον διορίσουμε αντιπρόεδρο. Ευχαριστώ πολύ. Muchas gracias. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Αν γίνεται δεκτή αυτή η υποψηφιότητα διαβοής, θέλετε κάποιος ή κάποια να ψηφίσουμε. Όχι λοιπόν, διαβοής εγκρίνεται. Συγχαίρουμε λοιπόν τον κύριο Πιμέντα Λόπες και ζητούμε να προσέλθει εδώ. Eh, Πολύ καλά. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τις ψηφοφορίες για σήμερα. Πρώτη έκθεση που θα ψηφίσουμε είναι η έκθεση της κυρίας Ρέντκε για την ισότητα των φύλων και στην ψηφιακή εποχή. Έχετε φαντάζομαι τις κάρτες για να ψηφίσετε όλοι στις συσκευές έτοιμες. Και ξεκινάμε λοιπόν με την ψηφοφορία. Τροπολογία 66 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 67 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 68. 68 καταπίπτει 68. 69 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 70 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε 71 αποσύρθηκε συμβιβασμός 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε προχωράμε στο συμβιβασμό 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε τροπολογία 81 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Τροπολογία 82 και 83 από κοινού αυτές υπέρ αυτών κατά αποχές εγκρίθηκαν. Τροπολογία 84 πίπτη. Η τροπολογία 86 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 87 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 88 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 89 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 93 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε Συμβιβασμός 16 υπέρ κατά απόχες εγκρίθηκε. Συμβιβασμός 17 υπέρ κατά απόχες εγκρίθηκε. Περνάμε στην τροπολογία 104-105 που είναι ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκαν. Συμβιβασμός 18 υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά ψηφίζουμε τη συμβιβαστική τροπολογία 18 άρχεται η ψηφοφορία υπάρχει κάποιος που δεν είμαστε τώρα πλήρης Πέρας ψηφοφορίας εγκρίθηκε η 18. Περνάμε στην σχόλιο χωρίς μικρόφωνο. Δεν ακούστηκε. Εντάξει, θα επαναλάβουμε λοιπόν την ψηφοφορία. Παρακαλώ να προσέχετε. Είπα ότι κάποιοι δεν ψήφισαν και στο τέλος έτσι παραμείναμε. Ψηφίζουμε την 18 ηλεκτρονικά. Άρχεται. Λοιπόν, να αναμείνουμε. Κάποιοι που δεν έχουν ψηφίσει. Πέρας ψηφοφορίας. Τώρα εντάξει πλέον. Απορρίφθηκε, απορρίφθηκε. Τροπολογία 42. Συγγνώμη, 92 υπέρ. 92. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε πάλι ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε την 92. Λοιπόν, να εστιαστούμε στην ψήφιση. Έλεγχος στις 92 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας απορρίφθηκε 106 τροπολογία υπέρ. Σε δύο τμήματα, συγγνώμη, ε, συγγνώμη, πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές Λοιπόν, θα ελέγξουμε τώρα πάλι το δεύτερο τμήμα της 106. Άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε το δεύτερο τμήμα. Τροπολογία 107 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 108 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίφθηκε. Συμβιβασμός 19 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. Συμβιβασμός 20 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 114 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 115 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 116 υπέρ για την 115 να ελέγξουμε λέτε εντάξει ψηφίζουμε ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία 115 Πέρας ψηφοφορίας. Σαφές. Δεν έκανα λάθος από ό,τι είδα. Έτσι απορρίφθηκε πράγματι. 116 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. 117 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 118 υπέρ. Όχι καταπίπτει, συγγνώμη, η 118 καταπίπτει επειδή η προηγούμενη εγκρίθηκε 119 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίφθηκε 120 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε της Επιτροπής Απασχόλησης 2 ΕΜΠΛ 2 δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε δεύτερο τμήμα υπέρ όχι, συγγνώμη, καλύπτεται το δεύτερο, δεν θα το ψηφίσουμε. 121 τροπολογία, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. 122 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. 123 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. 124 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. της απασχόλησης 12, έμπλ 12 καταπίπτει. Έτσι. Επειδή εγκρίθηκε η 123. Συμβιβασμός 21 υπέρ κατά απόχες εγκρίθηκε. Συμβιβασμός όχι, συγγνώμη. Τροπολογία 130 υπέρ κατά απόχες εγκρίθηκε. Έμπλ 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 131 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 132 υπέρ ...132 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Έμπρε 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έμπρε 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Έμπρε 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Έμπρε 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 134-135 ταυτόσημες υπέρ αυτών κατά αποχές απορρίφθηκαν 136 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 137 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 138 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 139 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε συμβαστική 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε περνάμε στην τροπολογία 142 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 143 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 144 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε συμβιβαστική 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε τροπολογία 147 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε να ελέγξουμε, θέλετε να ελέγξουμε αυτήν. Εντάξει, ελέγχουμε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 147. Άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. 149 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίφθηκε. 150 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίφθηκε. 151 αποσύρθηκε. 152 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 153 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 154 και 11 είναι ταυτόσιμες υπέρ αυτών κατά αποχές εγκρίθηκαν 155 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 156 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε Έμπλ 19. Πρώτο τμήμα δεν θα ψηφιστεί, διότι καλύπτεται ήδη. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Έμπλ 23, πρώτο τμήμα, δεν θα ψηφιστεί. Δεύτερο τμήμα θα ψηφίσουμε υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Τροπολογία 157, 158 και 159 ταυτόσημες υπέρ αυτών. Κατά αποχές απορρίφθηκαν. 160 υπέρ. Ε, κατά αποχές απορρίφθηκε. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε την 160. Άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Όχι ότι είχα δει αυτό το αποτέλεσμα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Δεν ξέρω, υπάρχουν, υπάρχει κάποια κάρτα που έχει μπει στη συσκευή και δεν ψηφίζει κάποιος. Εν πάση περιπτώσει, αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, τι να κάνουμε. Περνάμε τώρα στην, μια στιγμή, 161, υπέρ, κατά, άποχες εγκρίθηκε 163 υπέρ κατά άποχες εγκρίθηκε συμβιβασμός 24 υπέρ κατά άποχες εγκρίθηκε τροπολογία 168 υπέρ κατά άποχες απορρίφθηκε 169 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 170 171 υπέρ αυτών κατά αποχές απορρίφθηκαν 172 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 173 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 174 175 υπέρ αυτών κατά αποχές απορρίφθηκαν 176 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 177 και 178 υπέρ αυτών κατά αποχές απορρίφθηκαν 179 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 180 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 181 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε περνάμε στη συμβιβαστική 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε πάμε στην τροπολογία 193 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε συμβαστική 26 υπέρ κατά αποχές. Νομίζω ότι εγκρίθηκε, αλλά δεν είμαι σίγουρη. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για να ελέγξουμε. Άρχεται, ψηφίζουμε την 26, συμβαστική. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Συμβαστική 27. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Τοπολογία 198 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 199 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 200 να ελέγξουμε την πια την 199 εντάξει άρχεται η ψηφοφορία ψηφίζουμε την 199 Ψηφίσατε όλοι. Υπάρχει ένας παραπάνω από το... Υπάρχει, λέω, από το ΕΛΚ. Έχετε μια ψήφο παραπάνω. Κάποιος ψηφίζει παραπάνω από το ΕΛΚ. Πρέπει να αφαιρεθεί κάποιος. Μια ψήφος. Όχι, τώρα εντάξει. Ωραία. Ας συνεχίσουμε. Λοιπόν, και πάλι τώρα το ξανακάνατε. Να συμφωνήσετε τι θα κάνετε τελικά. Απορρίφθηκε λοιπόν. Τροπολογία 200 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 201 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. 201 να ελέγξουμε. Εντάξει ψηφίζουμε την 201. Άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας απορρίφθηκε για, με δύο ψήφους διαφορά. 202 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε πάλι λοιπόν. Ψηφίζουμε την 202 άρχεται η ψηφοφορία. Πάλι ένας παραπάνω ψηφίζει από το ΕΛΚ. Εντάξει τώρα πέρας ψηφοφορίας και αποτέλεσμα εγκρίθηκε. Συμβιβαστική 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Πάμε στην τροπολογία 208 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 209 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 211 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 212 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 213 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 214 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε συμβιβασμός 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε Θέλετε να ελέγξουμε για τη συμβαστική 29. Ναι, εντάξει να το κάνουμε. Αλλά εγώ βλέπω τις ομάδες πάνω κάτω πώς ψηφίζουν, αλλά εντάξει υπάρχουν κάποιοι που δεν σηκώνουν το χέρι. Ελέγχουμε λοιπόν, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά τη συμβαστική 29. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίθηκε συμβιβαστική 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε τροπολογία 217 υπέρ κατά αποχές δεν είδα σαφές το αποτέλεσμα ελέγχουμε ψηφίζουμε την 217 άρχεται η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας και αποτέλεσμα εγκρίθηκε Συμβιβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 15 υπέρ. Όχι, κάτι ξέχασα. Ναι, συμβιβαστική 2, συγγνώμη, ναι, συμβιβαστική 2 υπέρ. Κατά απόχες εγκρίθηκε. Τώρα ναι, η 15 υπέρ. Κατά απόχες εγκρίθηκε. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε συμβιβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε Προπολογία 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε συμβιβαστική συμβιβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε Συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 31 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 33 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 34 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Συμβιβαστική 7 υπέρ κατά αποχές Συμβιβαστική 7 θα ελέγξουμε. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται. Ψηφίζουμε τη συμβαστική 7. Εγκρίθηκε. Συμβιβασμός 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Συμβιβαστική 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Έμπρ σε υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε συμβιβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε τροπολογία 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε συμβιβασμός 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε τροπολογία 49 υπέρ ναι μετά τον συμβιβασμό περνάμε στην 49. 49 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. 50 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. 51 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. 52 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. 53 υπέρ, κατά αποχές δεν είναι σαφές θα ελέγξουμε ψηφίζουμε την 53 άρχεται πέρας ψηφοφορίας εγκρίθηκε 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 56 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε συμβαστική 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε τοπολογία 60 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 64 υπέρ κατά απόχέ εγκρίθηκε στην 2 τώρα τροπολογία υπέρ κατά απόχέ, απορρίφθηκε 3 υπέρ κατά απόχέ, απορρίφθηκε 4 υπέρ κατά Αποχέ. εγκρίθηκε 5 υπέρ κατά Αποχέ, απορρίφθηκε 6 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε έμπρ αιτιολογική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε έμπρ 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε έμπρ 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 1 δεν γίνεται αποδεκτή. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά το σύνολο της έκθεσης όπως τροποποιήθηκε. Άρχεται η ψηφοφορία. Ε, δεν πειράζει. Τι να κάνουμε. Ε. Ένας παραπάνω από το ΕΛΚ. Το ΕΛΚΑ έχει έναν που ψηφίζει και είναι επιπλέον. Λοιπόν τώρα εντάξει. Λοιπόν. Οκ. Okay. Να μην αφαιρεθούν άλλοι. Πολύ καλά. Εγκρίθηκε η έκθεση με 24 ψήφους υπέρ, 6 εναντίον, μία αποχή. Συγχαρητήρια λοιπόν στην εισηγήτρια. Vale, Εντάξει, ωραία, ελάτε, περνάμε τώρα. Ας προχωρήσουμε γρήγορα γιατί δεν έχουμε ξεκινήσει. Ε, έχουμε τώρα βρεθήκαμε με ορμή και έχουμε ένα καλό ρυθμό, συνεχίσουμε. Έχουμε το mainstreaming, την ένταξη της ισότητας των φίλων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τη κυρία Μίρνερ είναι η συγγήτρα. Είχαμε χθε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θα ψηφίσουμε την έκθεση αυτή σήμερα. Τροπολογία 45 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. 46 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 47 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. Συμβιβασμός 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 50 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. 51 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε συμβασμός 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε τροπολογία 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 57 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 58 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 59 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε έχουμε μια προφορική τροποποίηση στην, στο εδάφιο 9 ή όχι α έχουμε την αρχική παράγραφο αρχική παράγραφο στις 9 το ΕΛΚ ζήτησε ξεχωριστή ψηφοφορία σε τμήματα. Πρώτο τμήμα λοιπόν της 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα της 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 60 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 61 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 62 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίφθηκε 64 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Περνάμε τώρα στην τροπολογία 67 με μια προφορική τροποποίηση εδώ. Υπάρχει κάποια αντίρρηση στην προφορική τροποποίηση ή όχι. Όχι. Ωραία, ψηφίζουμε. 67 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 68 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε συμβασμός 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε συμβασμός 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε τροπολογία 77 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 78 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 79 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι απορρίφθηκε αλλά δεν είμαι σίγουρη θα ελέγξουμε λοιπόν την 79 ψηφίζουμε άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά πέρας ψηφοφορίας και αποτέλεσμα εγκρίθηκε. Τροπολογία 80 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 81 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 82 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 83 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 84 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε τροπολογία 91 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 93 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 94 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 95 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 96 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 100 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε πάμε στην τροπολογία 108 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 110 υπέρ κατά αποχές αεγκρίθηκε 109 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 113 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 114 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές δεν είμαι σίγουρη. Λοιπόν, ο συμβιβασμός 9 εγκρίθηκε. Εντάξει, 118 τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. 119 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. 120 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. 121 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. 122 υπέρ,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 κατά αποχές εγκρίθηκε 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 3 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 4 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε εγκρίθηκε συγγνώμη εγκρίθηκε 5 υπέρ 5 και 6 υπέρ αυτών κατά αποχές εγκρίθηκαν 7 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 12 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 11 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για να ελέγξουμε την 11 άρχεται Ήταν σαφές λοιπόν, απορρίφθηκε μάλιστα. Τροπολογία 13, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίθηκε. 14, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε 15 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε Ποια λέτε, τη 18. Ναι, είπα εγκρίθηκε ενώ απορρίφθηκε. Εντάξει, σωστό. Απορρίφθηκε, ναι, εντάξει. Αν θέλετε να το ελέγξουμε, εντάξει, ήταν σαφές όμως. Τροπολογία 19, υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίφθηκε. 20, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίθηκε. 21, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίθηκε 22 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 23 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 24 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 27 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 29 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 33 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 34 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε πάμε στην τροπολογία 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 44 υπέρ υπέρ της 44 κατά αποχές εγκρίθηκε και τώρα θα ψηφίσουμε στην έκθεση συνολικά άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίθηκε με 23 ψήφους υπέρ 6 κατά και μία αποχή. Συγχαρητήρια κυρία Μίρναρ. Και περνάμε στην ψήφιση της επόμενης έκθεσης ε, για τις γυναίκες που απασχολούνται το οικιακές βοηθοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση της κυρίας Κούνεβα. Ξεκινάμε με την ψηφοφορία. Συμβιβασμός 1 υπέρ. Κατά. Να δούμε λοιπόν μια στιγμή να επικεντρωθούμε σωστά στην ψηφοφορία. Συμβιβασμός 1 λοιπόν υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι εγκρίθηκε αλλά θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά ψηφίζουμε τη συμβαστική 1 άρχεται πέρας ψηφοφορίας εγκρίθηκε περνάμε στον συμβασμό 2 υπέρ κατά Μάλιστα. Λοιπόν, παρακαλώ πολύ. Ψηφίζουμε. Δεν βλέπω περισσότερους από αυτούς που σηκώνουν τα χέρια. Αν δεν σηκώνετε τα χέρια τι να κάνουμε. Όχι μόνο υπάρχει και η κακή διάθεση αλλά αρχίζω και εξοργίζομαι στο τέλος με αυτή την κατάσταση. Εν πάση περιπτώσει, συμβιβασμός 2 υπέρ λοιπόν. Κατά αποχές, νομίζω απορρίφθηκε, απορρίφθηκε ναι. Γι' αυτό λοιπόν να ελέγξουμε, ωραία. Ψηφίζουμε το συμβασμό 2, άρχεται η ψηφοφορία. Να κλείσουμε τώρα. Προσέξτε, για δείτε τι έγινε. Μάλιστα, εγκρίθηκε η συμβαστική 2. Εγκρίθηκε. Πάμε λοιπόν στην 83 τροπολογία. Υπέρ. Κατά αποχές. Κανείς δεν ψηφίζει. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, τι γίνεται εδώ. Περί τίνος πρόκειται. Λοιπόν, τροπολογία 83 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε την 83. Άρχεται. πέρας ψηφοφορίας εγκρίθηκε συμβιβασμός 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε τροπολογία 89 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 148 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε Συμβιβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 98 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 93 και 94 είναι ταυτόσιμες υπέρ αυτών. Κατά. Αποχές. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά την 94. Άρχεται η ψηφοφορία. εγκρίθηκε. Είναι προφανές έτσι, αλλά αν σηκώνουμε τα χέρια δεν θα χρειαζόταν ηλεκτρονική επαλήθευση. Τέλος πάντων, 94 εγκρίθηκε, 95 τώρα. Όχι, καταπίπτει, μια και εγκρίθηκε η άλλη. 96 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. 97 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. 99 υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε 100 αποσύρθηκε 100 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 101 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 103 υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε ψηφίζουμε την 103 άρχεται Πέρας ψηφοφορία. Εγκρίθηκε. Πάμε λοιπόν τώρα στην συμβαστική 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 112. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. 111. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκε 114 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 115 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 113 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 152 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 116 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 117 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά, ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα της 117. Άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε έμπλ 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε καταπίπτει αυτή η 118 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 123 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 119 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 120 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 121 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 122 υπέρ κατά ε, αποχές εγκρίθηκε 129 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 124 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε Συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 128 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 130 υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε ψηφίζουμε την 130 ηλεκτρονικά άρχεται Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. 131 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. 132 υπέρ. Να ελέγξουμε λέτε την 131. Ωραία. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Λοιπόν, είχατε δίκιο. Με μία ψήφο διαφορά εγκρίθηκε. Πράγματι είχατε δίκιο. Ωραία. 132 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίφθηκε. Η 107. Μόνο το δεύτερο τμήμα της. Ψηφίζουμε υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Έμπλη 22 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε τροπολογία 134 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 136 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 137 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 138 υπέρ με μια προφορική τροποποίηση που εντάσσεται στο κείμενο η προφορική τροποποίηση. Αποσύρω την τροπολογία. Πληροφορική τροπολογία. Πολύ καλά, πολύ καλά. Με την προφορική τροπολογία που αποσύρθηκε ψηφίζουμε λοιπόν την 138 ως έχει. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκε 109 υπέρ λοιπόν ήταν προφανές ναι 109 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε έμπλ 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε Έμπλουτρια υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε τροπολογία 163 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 149 υπέρ όχι καταπίπτει επειδή εγκρίθηκε η 163 συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 110 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 150 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 139 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε έμπλη 23 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε τροπολογία 133 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 151 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 153 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 154 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 155 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 156 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 157 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Έμπλου 40 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Έμπλου 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 162 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 164 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 165 υπέρ κατά αποχές 165 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε παρακαλώ σηκώντε τα χέρια σας γιατί διαφορετικά δεν μπορούμε να δούμε τι γίνεται έμπλ 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε έμπλ 19 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε έμπλ 25 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε έμπλ 26 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε έμπλη 28 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε έμπλη 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε έμπλη 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε έμπλη 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε έμπλη 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε MP35 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε MP37 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε MP42 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε το υπόλοιπο Τη Σέμπλ δεν θα ψηφιστεί. Πολύ καλό αυτό, ε. Ωραία. Τροπολογία 1 τώρα, υπέρ. Κατά. Λοιπόν, προσοχή. Τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 4 και 6 υπέρ αυτών κατά αποχές εγκρίθηκαν. 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε η 8 καταπίπτει η 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 10 καταπίπτει 25 επίσης 26 τώρα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε Ψηφίζεται αυτή έτσι. Έμπλ 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 21 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 19 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 12 υπέρ συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε H υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε W υπέρ κατά υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται να ελέγξουμε ελέγχουμε λοιπόν την W άρχεται η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας είχατε δίκιο απορρίφθηκε Προπολογία 28 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 30 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 31 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Η 33 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. Να ελέγξουμε για το δεύτερο τμήμα. Εντάξει, ελέγχουμε. Ψηφίζουμε την 33 δεύτερο τμήμα. Άρχεται. Απορρίφθηκε. Συμβαστική 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Συμβαστική 14. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε έμπλ α ε, υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε Emperor T υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε συμβαστική 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβιβαστική 16 υπέρ κατά αποχές. Δεν είναι σαφές. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για επαλήθευση. Ψηφίζουμε τη συμβαστική 16. Απορρίφθηκε. Και έτσι πάμε στην 44 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 45 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 46 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 48 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Προσοχή. Δεν εγκρίθηκε ο συμβιβασμός 16. Πρέπει να ψηφίσουμε όλες τις τροπολογίες λοιπόν. Τώρα ψηφίζουμε τις 48 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα λοιπόν υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Έλεγχος. Ωραία. Θα ψηφίσουμε το δεύτερο τμήμα ηλεκτρονικά τις 48. Άρχεται. Δεύτερο τμήμα. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίθηκε λοιπόν. Μάλιστα. 47. Όχι, όχι, συγγνώμη. Έμπλ 6 πρώτα. Έμπλ 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Τώρα η 47 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 49 υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκε 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 52 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε συμβαστική 17 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε Τοπολογία 64 υπέρ 54 με συγχωρείτε υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε έμπλ 5 ρωμαϊκό β υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 65 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 55 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 29 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε Q υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε AG υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε πάμε στην 59 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε έμπερ υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε έμπλ AM υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε συμβαστική 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε συμβαστική 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε έμπλ AL υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε τροπολογία 62 χωρίς μικρόφωνο. Μάλιστα, ψηφίζουμε την 62 τώρα. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Συμβιβαστική 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Έμπρ Z υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε την Emperor Z. Άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίθηκε. Ήταν προφανέστατο με το αποτέλεσμα αυτό εγκρίθηκε. ΕΚ AK υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 68 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 69 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε τροπολογία 70 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε συμβαστική 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 72 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε συμβαστική 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε συμβαστική 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε Emperor D υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε Emperor F υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε L υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε M υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε N υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε AB υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε AC υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε AD υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε AE υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε AF υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Και περνάμε τώρα στην τελική ηλεκτρονική ψήφιση. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά, παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας και εγκρίθηκε με 16 ψήφους υπέρ, μία εναντίον και 14 αποχές. Συγχαρητήρια κυρία Κούνεβα. Λοιπόν, προχωράμε. Δεν απομένει πια τίποτα. Αυτή η τελευταία είναι πολύ πιο ελαφριά αυτή η έκθεση. Είναι η πρώτη τελευταία όμως, ε, ναι. Ωραία. Εντάξει, ούτε και η τελευταία όμως είναι μεγάλη. Ψηφίζουμε λοιπόν την έκθεση για την εφαρμογή της οδηγίας για την γονική άδεια, parental leave, η συγγήτρια, εγώ ίδια, η κυρία Γκαρθία Πέρεθ και περνάμε και ψηφίζουμε κατευθείαν. Συμβιβαστική 1 υπέρ κατά αποχές. Λοιπόν, προσοχή, ηλεκτρονική, ηλεκτρονικός έλεγχος, συμβαστική 1, άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 20 υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκε για την 20 να ελέγξουμε να ελέγξουμε την 20 έτσι ωραία άρχεται απορρίφθηκε 21 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 23 αποσύρθηκε. Συμβιβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Νομίζω, εντάξει, να ελέγξουμε. Ψηφίζουμε συμβιβαστική 2 άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε, απορρίφθηκε, μάλιστα. Συνεχίζουμε λοιπόν 24 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 25 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 27 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε ψηφίζουμε το δεύτερο τμήμα της 27 άρχεται πέρας ψηφοφορίας απορρίφθηκε 28 αποσύρθηκε συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε τροπολογία 30 με μια προφορική τροποποίηση που την έχετε στα χαρτιά σας στο κείμενο ψηφίζουμε την 30 ως έχει με την τροποποίηση υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 34 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 35 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε Ε, τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε Τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 2 υπέρ χωρίς μικρόφωνο. Η τροπολογία 2 λοιπόν υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 4 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε Σύμβασ... Α, η έξι πρώτα, συγγνώμη, υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 13 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίφθηκε, απορρίφθηκε, συγγνώμη, συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές. Νομίζω απορρίφθηκε, αλλά θα ελέγξουμε. Άρχεται, ψηφίζουμε τη συμβαστική 6. Υπάρχουν κάποιοι που ή δεν θέλουν να ψηφίσουν ή τι γίνεται με την κάρτα τους. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ελάτε τώρα. Ρετσαθάδα. Απορρίφθηκε, απορρίφθηκε ο συμβιβασμός. 14 τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Τροπολογία 15 υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε η 16 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε και περνάμε και ψηφίζουμε τώρα σε τελική ψηφοφορία την έκθεση άρχεται και εγκρίθηκε με 17 ψήφους υπέρ, 13 εναντίον, μία αποχή. Εκείνη, αφού είναι δική της η έκθεση, συγχαίρω τον εαυτό μου. Λοιπόν, η τελευταία τώρα έκθεση που ψηφίζουμε για το κοινωνικό dumping στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η συγγήτρια η κυρία Ρέγνερ. Ξεκινάμε με την ψηφοφορία. Συμβαστική 3, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Τροπολογία 20, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. 21, υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 22 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε τροπολογία 23 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 25 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 26 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 27 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 28 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε πάμε στην τροπολογία 35 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 36 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 37 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 39 καταπίπτει 39 συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Πάμε στην τροπολογία 45 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 47 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 48 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 49 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 50 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 51 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 52 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 53 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε Τοπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές εγ... όχι τροπολογία 4 λοιπόν υπέρ ξανά αποχές, κατά αποχές απορρίφθηκε. Τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Η 7 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Η 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 11 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 13 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε τελική ψηφοφορία τώρα άρχεται η ψηφοφορία εγκρίθηκε η έκθεση με 28 ψήφους υπέρ, μία εναντίον και δύο αποχές. Συγχαρητήρια κυρία Ρέγνερ. Και έληξε εδώ, ολοκληρώθηκε το έργο της Επιτροπής μας. Ευχαριστώ για τη συνεργασία σας. Να περάσετε μια καλή εβδομάδα, υπόλοιπο εβδομάδα. Γεια σας.